Παρακαλώ, κύριε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, παίρνω το λόγο για να σας πω ότι η ομάδα των κομμουνιστών ε, δεν συμμετείχαν στην τελετή. Αυτή ο μη σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι όνειδος. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ίσως μπορείτε να πείτε ότι σήμερα το πρωί, αύριο το πρωί θα έχουμε, ε, θα πρέπει ε, να συγχαρούμε ε, τις, τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά για τον τρόπο των εκλογών. Η Σομαλία, Σομαλία έχει δεσμευτεί στην δημοκρατία στο κράτος δικαίου και θα έπρεπε να γίνει ένα κράτος πλήρως ανεγνωρισμένο και να γίνει δεκτό στην οικογένεια των εθνών. Η Σομαλιλάνδη. Ευχαριστούμε πριν από την ψηφοφορία ήθελα να εκφράσω την ανησυχία μας για τον καθηγητή ερευνητή από το Ελευθερή, από το Ελεύθερο Πανεπιστημίο ε, των Βρυξελών, η οποία μάλλον ε, καταδικάστηκε από τι Αρχές με την κατηγορία της κατασκοπίας. Η επιστολή μου προς τον πρόεδρο της χώρας, όπου ζητώ την απελευθέρωση της ε, κυρίας Γελάρη, είναι και μια δίκαιη δίκη δεν έχει λάβει απάντηση προς στιγμή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρός κινδύνος, κυρία Νταλάρη, να ε,